Ladies Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας που συνδυάζει σήμερα και αύριο. Καταρχήν να μου πείτε αν έχετε παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε εσείς προτάσεις αλλαγή της ημερήσιας διάταξης, θα σας πω εγώ τι τροποποιήσεις υπάρχουν. Για τη διερμηνία είχαμε κάποια προβλήματα με τα ρουμανικά, αλλά νομίζω ότι έχουν ρυθμιστεί τα, τα προβλήματα. Ε, να σας πω ότι ο εισηγητής ε, για το ΕΝΙΖΑ, ο κ. Τσίτσεστερ, έχει προτείνει την ε, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου ως ημερομηνία για την ψηφοφορία για την έκθεση ΕΝΙΖΑ. Ε, θα θέλω επίσης να καλωσορίσουμε κάποια νέα μέλη. Δεν είναι όλα τα νέα μέλη, αλλά αν είναι κάποιοι εδώ, σηκωθούν παρακαλώ, ας εγερθούν τα νέα μέλη. Ο κύριος Γκιούρκ, δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Ο κύριος Σαλβαδός εδώ, η Αλαμπάρτ. Επίσης δεν είναι εδώ. Αντρέ Μπαρέα. Αμέλια Ντότερ, Λορέντζο Φοντάνα. Και νέοι αναπληρωτές. Σοφία Ματσέγη Κούκοβιτς. Ζαν Ροάτα και Τζίνο Τρεματέρα. Έχουμε λοιπόν νέα μέλη στην Επιτροπή μας. όπως αποφασίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων. Έχουμε επομένω επιπλέον μέλη στην Επιτροπή μας, αλλά δεν είχαν χρόνο σήμερα για να έρθουν, οπότε είμαστε σε αρκετά περιορισμένη ε, σύνθεση. Θα πρέπει επίσης να σας ανακοινώσω μία μίνι ακρόαση ο κύριος Βίνιε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαλειτουργικών Συστημάτων έχει αντικατασταθεί από την κυρία Ανδριανή Φέρτη και ο Πολωνός Υπουργός για την ακρόαση είναι ο Υπουργός κύριος Ιγκόρ Οστρόφσκι, Υφυπουργός στο Υπουργείο Διοίκησης και Ψηφιοποίησης. Και στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης ο αναπληρωτής Πρωθυπουργό και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται, δεν θα έρθει ο κύριος Πόλακ, αλλά θα έρθει ο καθηγητής κύριος Μάτσιακ Καλίσκι. Και στο σημείο 13, πάλι μια αντικατάσταση, θα έχουμε την Υπουργό Μαγκαλένα Γκάλι, αντικαθιστώντας τον Πολωνό Υπουργό Μίχαελ Μπόνι. Αρκετές λοιπόν αλλαγές και αντικαταστάσεις. Τώρα όμως σας τα ανακοίνωσα και αν δεν έχετε αντιρρήσει αυτή είναι η ημερήσια διάταξη, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Περνάμε στο πρώτο σημείο για τη σημερινή ημερήσια διάταξη, αφού θέλουμε να προχωρήσουμε και σχετικά γρήγορα για να μας μείνει χρόνος για τη συζήτηση. Αναθεώρηση του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το έβδομο ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Έχουμε γνωμοδότηση και υπεύθυνη συντάκτρια είναι η κυρία Κριστίνα Γκουτιέρες Κορτίνες και σας δίνουμε το λόγο και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές και ενδιαφερομένους συναδέλφους, αλλά ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι σήμερα δεν είναι και πάρα πολλοί εδώ. Κυρία συνάδελφα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την έκθεση, αν και είναι απλώ μια γνωμοδότηση, αλλά εγώ ήμουν και το 2002 εισηγήτρια για αυτό το ίδιο πρόγραμμα για το περιβάλλον και μπορώ να κάνω μια σύγκριση μεταξύ αυτού που συνέβη τότε και του τι συμβαίνει τώρα. Και ήθελα να πω κάτι που μου φαίνεται σημαντικό η δομή και οι αρμοδιότητες ε, της γενική Διεύθυνσης, της Γενική Επιτροπή για το Περιβάλλον περιορίστηκαν πάρα πολύ από τότε. Έχουμε ενώπιον μα άλλη Γενική Διεύθυνση με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και, ε, αν, ε, και επίσης ε, αφαιρέθηκα από τις αρμοδιότητες της η κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι πολλοί σε αυτό τον οίκο βέβαια δεν το κατάλαβαν. Έτσι λοιπόν δίνουν σε αυτό το φορέα αρμοδιότητες που δεν έχει. Τώρα ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχει εγώ. Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να το παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι η βιοπικιλότητα είναι ε, ουσιαστικά το πιο σημαντικό και έχουμε μέσα σε αρμοδιότητες όλα όσα έχουν να κάνουν με τη βιοπικιλότητα αλλά ποτέ δεν ε, είναι αρκετά προσδιορισμένο. Έχουμε την ε, διατήρηση του εδάφους, την προστασία των οικοσυστημάτων, το θέμα του ύδατος και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φέτος έχουμε το blueprint για το είδωρ και έχουμε ε, επίσης και ένα άλλο πρόγραμμα ε, για το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η ίδια Γενική Διεύθυνση δεν ε, αντέδρασε προ το στρόκ να μείνει χωρί κλιματική αλλαγή. Γιατί, αν και είναι κάτι πολύ διαδεδομένο το θέμα τη κλιματική αλλαγή, είναι ένας ε, παράγοντας που θα προσέδιδε μεγάλη ισχύ σε αυτό το φορέα, ενώ οι υπόλοιπε παρουσιάστηκαν ως συγκεκριμένε πολιτικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένε πολιτικές, η βιοπικιλότητα κτλ. Όμω, ουσιαστικά, προσπάθησαν εδώ να, δοθούν, να δοθεί έμφυση ε, στα προβλήματα που μπορούν να αφορούν το Κοινοβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι όλα όσα λέγονται είναι πολύ γενικόλογα και δεν υπάρχει καμία δέσμευση και θα έλεγα ότι ο λόγος είναι πολύ θεωρητικός και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε ακόμη και αν το λες στην έκθεση είναι πώς ε, θα ληφθούν τα μέτρα και πώς θα εφαρμοστούν προκειμένου ε, ο εν λόγω φορέας ε, να μπορέσει να υλοποιήσει τις ε, αρμοδιότητες που έχει αναλάβει. Ακόμη και με φαντασία θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί διαφορετικό θέμα είναι οι αρμοδιότητες και διαφορετικό είναι το να εμφανίζει κάποια ηγετική θέση. αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε να εμφανίσει ηγετική θέση, γιατί ένα από τα κύρια θέματα που τέθηκαν στην πρώτη γραμμή είναι το θέμα του πόσο σημαντική είναι στην καθημερινή ζωή ο αντίκτυπο τη οδηγία που αναθεωρήθηκε το 2002. Όλα τα διαφορετικά ταμεία, όλα τα μεγάλα έργα, όλα εξαρτώνται από την οδηγία για τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και όλα είναι γίνεται και πιο ισχυρή και πιο ενισχυμένη. Και παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η διαχείρισή τη δεν είναι καλή γιατί η οδηγία επικεντρώθηκε στην ε, πράξη σε ένα τμήμα των όσων ε, πρέπει να τρεπασχολούν. Δηλαδή, ο αντίκτυπος ε, στην φύση, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπο στο έδαφο, ε, στην ιστορική κληρονομιά, ο αντίκτυπο τη πόλη, ε, στο τοπίο. Γι' αυτό υπάρχει στο διατακτικό, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το ελέγχει. Στην Επιτροπή Αναφορών είχαμε πάρα πολλέ αιτήσει που υπάρχει, παραδείγματο χάρη, ένα δρόμο που περνάει από ε, ένα ιστορικό αρχαιολογικό χώρο και δεν έλειφθη υπόψη για το σχεδιασμό του αυτοκινητόδρομου όμως. Στη μεγαλύτερη περίπτωση ε, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών είναι βιολόγοι, βιτονολόγοι και παραδείγματος χάρη ε, δεν έχουν καμία σχέση παραδείγματο χάρη με ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή, αν περνάει ο αυτοκινητόδρομο σε ένα μέρο όπου κατοίκησαν οι πρώτοι βασιλιάδε στην Ιρλανδία. Έτσι λοιπόν έχουμε τα θεωρητικά ζητήματα και το θέμα της συμβατότητας. Συμβατότητα των νεώσιμων πηγών ενέργειας με το τοπίο παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι ένα θέμα όπου θα έπρεπε να έχουμε ξεκάθαρες διατάξεις στην οδηγία. Και το ίδιο έχει να κάνει με το πού τοποθετούμε την ενέργεια. Θα πρέπει ε, να τα δούμε τα θέματα αυτά, αλλά από εκεί μέχρι να το βλέπουμε μηχανιστικά την οδηγία υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι λοιπόν ζητώ να ληφθεί υπόψη η ο, αναθεώρηση της οδηγίας για τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και σε όλες τις συνιστώσεις της. Ε, Παραδείγματο χάρη για το θέμα του τοπίου πριν 10 χρόνια ήταν λιγότερο σημαντικό αυτό το θέμα ε, από όσο σήμερα. Έχουμε και θέμα αισθητικής ε, και επίσης και για λόγους τουρισμού θέλουμε να έχουμε ένα όμορφο τοπίο. Δεύτερο θέμα, χρηματοδότηση από το Natura 2000. Μία από τις μεγάλες αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, το εξή. Εμεί θέλαμε ότι η Natura 2000 να προστατεύει και ε, λένε κάποιοι έχω το 20% το 40% του εδάφου μου που προστατεύεται όμω. Πώ γίνεται η διαχείριση, Γιατί πολλέ φορέ κάποιο θεωρεί ότι η προστασία είναι να μην κάνει τίποτα. Παραδείγματο χάρη ε, η έρημη επικράτεια. Ε, δηλαδή κανεί δεν μπορεί να μπει εκεί και δεν συμβαίνει τίποτα και ούτε καν παραγωγική είναι η γη. Έτσι λοιπόν για μένα η εφαρμογή της Natura 2000 και το άρθρο 6 δεν γίνεται σωστά γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη ότι τα ζώα ζουν από την ε, Γεωργία και κάτι πίνουν και κάτι τρώνε. το χάρη στην Νότια Ισπανία οι κυνηγοί ε, βάζουν ε, νερό, τοποθετούν νερό για να πάνε εκεί τα πουλιά, γιατί διαφορετικά δεν πάνε. Και ε, έχουμε ε, πάρα πολλές ε, περιπτώσεις όπου ε, διατηρείται σε ορισμένα αγροτεμάχια το σιτάρι για να πάνε να φάνε τα πουλιά και έχουμε παραδείγματο χάρη ε, επαρκή γεωργία για να στηρίξουμε τα οικοσυστήματα, όχι. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι τα σχέδια διαχείρισης της Natura 2000 δεν πρέπει να σημαίνουν απαγόρευση, αλλά συμφωνίες με τους stakeholders, με τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να γίνεται μια ορθή διαχείριση και να μπορεί να είναι και παραγωγικό το έδαφος με ένα συμβατό τρόπο. Και έχουμε και ορισμένους ε, που θέλουν να αγοράσουν προστατευόμενα εδάφη, όμως πρέπει ε, αυτός που θα είναι διοκτήτης να είναι και κυπουρός κατά κάποιο τρόπο ε, αυτής της επικράτειας. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πρόγραμμα για την εφαρμογή και όχι μόνο με απαγόρευση. Και επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα της ρύθμισης ε, του εδάφους. Εγώ Θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένη η οδηγία για την προστασία του εδάφους. Ε, υπάρχουν ε, κάποια ελάχιστα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, που είναι το δικαίωμα των πολιτών για να ξέρουν πού είναι τα μολυσμένα εδάφη ή ορισμένα κριτήρια για το πώς και πού κατασκευάζονται αυτοκινητόδρομοι γιατί πολλές από τις πλημμύρες που έχουμε οφείλονται στο ότι έχουμε αυτοκινητόδρομους ε, που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε ρεματιές παραδείγματος χάρη. Έτσι λοιπόν, για να αποφύγουμε τις κατολιστήσει και τις καταστροφές και τις τραγωδίες και πολλές φορές πλημμύρες, πρέπει να έχουμε τα ελάχιστα κριτήρια για την ε, διατήρηση και την προστασία του εδάφους. Γιατί, παραδείγματο χάρη, ε, στη Γαλλία μιλάμε ε, για το ότι το έδαφος μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο προορισμό. Δηλαδή, κάπου δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε σπίτια σε συγκεκριμένο έδαφο. Τώρα, από την άλλη. Νομίζω ότι μέχρι το 2050 πρέπει να δούμε τα προβλήματα καθολικά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια οδηγία για τα προστοκτόνα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το κλίμα. Εμείς στο Νότο ε, Παραδείγματο χάρη ε, παραπονιόμαστε γιατί όλη η οδηγία για τα παρασιτοκτόνα έχει να κάνει με του μήκητε. ενώ εμεί έχουμε έντομα εκεί, έχουμε κουρούπια πρέπει να λαμβάνονται και αυτά υπόψη, είναι εμεί. Δούμε ένα χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαφοροποιείται η Μεσόγειος από την ε, βόρεια περιοχή γιατί βλέπουμε διαφορετικά κλίμακα. Και αυτή η παλιά ιδέα ότι όλοι πρέπει να έχουμε το ίδιο κουστούμι ε, νομίζω Νομίζω ότι είναι μια αναποτελεσματική ιδέα και παλιωμοδίτικη. Ορισμένε φορέ πρέπει να προσαρμόζουμε τι οδηγίε στι συγκεκριμένε κλιματικέ συνθήκε των συγκεκριμένων περιοχών, γιατί διαφέρει το κλίμα και έχουμε διαφορετικέ συνθήκε και διαφορετικά προβλήματα. Και εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι σημαντικό για το πρόγραμμα LIFE. Εγώ ήμουν εισηγήτρια και για το LIFE. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ότι υπήρχε πραγματική επανάσταση στην περίπτωση των γυναικών. Ήμασταν πέντε γυναίκες ε, εισηγήτριε ε, για το LIFE και ξέρετε το LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο, εκτό από το κεφάλαιο 1, δηλαδή το μισθό των υπαλλήλων, τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το LIFE, χρηματοδότηση των προγραμμάτων, των ενισχύσεων, τα πάντα. Όμω το LIFE έχει και ένα τμήμα που αφορά τα προγράμματα, projects. Εμείς ε, κάναμε την πρώτη ανάγνωση στο live ε, και όταν ε, φτάσαμε στα κονδύλια ζήτησε κάποια χώρα να γίνει εθνικοποίηση του live, δηλαδή κάθε χώρα έπρεπε να επιλέξει τα προγράμματά της. Έτσι λοιπόν έγινε επανάσταση από την εισηγήτρια που ήταν στους Πρασίνους και από την κυρία Ινμαν από του σοσιαλιστέ και από μένα και αρνηθήκαμε. Βάλαμε μια τροπολογία και είπαμε ότι πρέπει να είναι ευρωπαϊκό το LIFE ω 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ή το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο ή το 6ο. Γιατί θέλαμε να εγγυηθούμε την ποιότητα και τα διεθνικά προγράμματα και τα δημαρχία ή ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει που ζητούν το live έπρεπε να το πράξουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει την επιλογή. Γιατί διαφορετικά επαναλαμβάνουμε την ίδια έρευνα και το ίδιο εγχείρημα ε, σε διάφορε χώρε. Τότε πληρώνει η Ευρώπη τέσσερι φορέ για το ίδιο πράγμα. Και είχαμε εκτό μήνε ε, για να ε, τον προπολογισμό της Κομισιόν. Τα καταφέραμε τελικά και ήταν θεαματικά τα αποτελέσματα του live και κατορθώσαμε το εξή. Ε, σήμερα έχουμε διεθνικά σχέδια γιατί όταν πετούν τα πουλιά παραδείγματο χάρη δεν ρωτάνε ε, ε, από ποια χώρα περνάνε όταν πηγαίνουν προς την Αφρική και όταν έχουμε προβλήματα κλιματικής αλλαγής ούτε παραδείγματος χάρη τα σύννεφα ρωτούν από ποια χώρα περνάνε. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδες το live να συνεχίζει να είναι διεθνές δηλαδή συνεργασία μεταξύ των χωρών και να αποφασίσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, θέλω να μιλήσω για το νερό. Πιστεύω ότι είχαμε ένα είδος ε, πολύ σκληρού φανταμεταλλισμού εναντί του νερού και ε, ξέρετε αυτή η οδηγία πλαίσιο για το είδωρ, ε, για το νερό είναι εξαιρετικό έγγραφο αλλά εκπροσωπεί ένα τμήμα δηλαδή πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των ποταμών, ε, των υπογείων υδάτων κατά την άποψή μου δεν είναι και τόσο καλή οδηγία αυτή για τα υπόγεια επιδέτα, αλλά έχουμε και το blueprint όπου γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα, έχουμε περισσότερες γνώσεις και εκεί πολλοί δήμοι και κράτη εφαρμόζουν ε, το κείμενο αυτό ε, για την ποιότητα του νερού πολύ αυστηρά και εκεί ε, και όπου έχουμε ε, αν δούμε ότι έχουμε την τεχνολογία για την ανακύκλωση του νερού και τη ανακύκλωση, τώρα πρέπει να μπούμε σε μια πιο επιστημονική και πολύπλοκη πολιτική για το νερό και να εργαστούμε χωρίς ε, προκαταλήψεις. Δηλαδή να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Όταν ε, μιλάμε για αφαλάτωση, πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς η ενέργεια καταναλώνεται και τι ρήπανση προκαλείται από την εγκατάσταση τη αφαλάτωση και μπορώ να σας πω ότι καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, πετάμε το αλάτι στη θάλασσα και καταστρέφεται όλη, ε, όλο το οικοσύστημα της θάλασσας. Πρέπει να υπάρχει αφαλάτωση, ναι, αλλά όχι ως η τέλεια λύση, εξαρτάται από το πού, από τον τόπο, γιατί η πρώτη αρχή της βιωσιμότητας είναι πού γίνονται τα πράγματα και με ποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια καθολική πολιτική για το υδρό. Αυτή την έκκληση επευθύνω στην Επιτροπή και να λαμβάνουμε υπόψη και την ανάκτηση του κύκλου του νερού. Δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη πώς γνωρίζουμε για τη βροχή, για τα ποτάμια, τη γνώση που έχουμε για τα θέματα αυτά και για την τεχνολογία. Και αυτό γιατί έχουμε κριτήρια, μέσα, χρήματα και κονδύλια για να ελέγξουμε τα τα παραδείγματος χάρη και Αυτά πρέπει να ελεγχθούν μεταξύ άλλων ε, γιατί ε, θα πρέπει να ελέγχουμε τους παράγοντες της ρήπασης και πρέπει να ξέρουμε πώς θα κάνουμε την αφαλάτωση, παραδείγματος χάρη. Νομίζω ότι η Γενική Διευθυνσή με αυτό το πρόγραμμα πρέπει να κάνει πάρα πολλά, αλλά πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά να εφαρμόσει όσα ε, γνωρίζει από την επιστήμη με πολύ σαφή τρόπο και να ακολουθήσει μια πιο επιστημονική προσέγγιση για την αναθεώρηση των οδηγιών. Πολλές φορές πρέπει να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συναδέλφε οι σκιώδεις συζητητές δεν είναι εδώ για να τους ρωτήσω αν θέλουν να πούν κάτι. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, μήπως θέλει να διευκρινίσει κάτι. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις ε, πολλές και χρήσιμες προτάσεις της. Ένα σημείο διευκρίνησης. Τα προγράμματα τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικά προγράμματα καθοδήγησης που μας βοηθούν να κρατήσουμε τον προσανατολισμό μας και στο τελευταίο πρόγραμμα είχαμε αρκετές αλλαγές. Ξεκινήσαμε από μια Ευρώπη 15 ε, κρατών μελών και έχουμε φτάσει σε μια Ευρώπη των 27 κρατών μελών. Επειδή ακριβώς υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές και επειδή το πρόγραμμα δράσης είχε πολλές αλλαγές κατά την υλοποίησή του. Ήταν σημαντικό ε, να εξηγήσουμε τι επέτυχε το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο πριν περάσουμε στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Και όπως είπε και η συγγήτρια, θέλουμε να επιτύχουμε. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει την απαραίτητη φαντασία που μας ζητάτε να δείξουμε. Και για να σχολιάσω λίγο αυτά τα οποία είπατε, Θέλω να πω ότι το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον θέλουμε ε, να εστιαστεί σε στόχους προτεραιότητας, θέλουμε ε, να αναλάβουν τα κράτη-μέλη δέσμευση σε μεγαλύτερο βαθμό για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα και να υλοποιήσουν ε, τις προτεραιότητες που θα ορίσει και το Κοινοβούλιο και αυτό το πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον θέλουμε να συνεισφέρει για τις πολιτικές και για την αποτελεσματικότητα των πόρων. Ορισμένα από τα ζητήματα που ανέφερε η συγγήτρια εδώ είναι πολύ σημαντικά, ιδίω τα θέματα των οικοσυστημάτων και τη προστασία του εδάφου, καθώ και το σημείο που ανέφερε για την προστασία των υδάτων. Θα ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, πράγμα το οποίο επιθυμεί και η συγγήτρια και ελπίζουμε ότι το 7ο πρόγραμμα δράσης θα μπορέσει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση. και στη γραπτή της γνωμοδότηση η συγγήτρια κάνει μια έκκληση σχετικά με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής για το Περιβάλλον, κάτι με το οποίο συμφωνούμε απολύτως όχι μόνο το πρόγραμμα LIFE, αλλά και άλλα προγράμματα χρειαζόμαστε και αυτό που είναι σημαντικό είναι το να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέργεια μεταξύ όλων αυτών των προγραμμάτων, ανταγωνιστικότητα, πρόγραμμα για τον ορίζοντα του 2020, πρόγραμμα ε, LIFE, θα συνεισφέρουν στην προστασία της βιοπικιλότητας και των εδαφών και των υδάτων. Για την τελευταία σας παρατήρηση σχετικά με τα υδάτα, το προσχέδιο θα εκδοθεί στο δεύτερο ήμιση του έτους και θα δώσει απαντήσεις σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Πώς μπορούμε να εντάξουμε την πολιτική για το νερό μέσα σε όλες τις άλλες πολιτικές και ε, με τον τρόπο θα να, έχουμε, να υποφεληθούμε από την υπάρχουσα γνώση για να τα κάνουμε όλα αυτά. Αναφέρετε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα για το νερό σε σχέση με την ε, αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άλλο που να θέλει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Κουτιέρη. Ξέχασα να πω κάτι και θα ήθελα να το πω για να είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτά που είπα. Η βιοπικιλότητα. Γιατί έχει αποτύχει μεταξύ άλλων η βιοπικιλότητα. Έχουμε επιλέξει έναν όρο που κανείς δεν τον καταλαβαίνει. Μπαίνω στο μετρό στη Μαδρίτη και ρωτάω Όποιο ξέρει τι θα πει ο να σηκώσει το χέρι. Κανείς δεν θα το σηκώσει. Γιατί ωραίο ακούγεται αλλά κανείς δεν ξέρει τι είναι. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Λένε οι μεγάλοι εμπειρογνώμες περιουσιάρι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν έντομα. Τα εξα... εξοντώνουμε. Και τα ζώα και τα πτηνά είναι άλλο ένα... Επίσης τα πουλιά εκλείπουν σιγά σιγά. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε συγκεκριμένες δράσεις. Μια παιδαγωγική εργασία την οποία δεν έχουμε κάνει ακόμη. Και θα ξεκινήσουμε και με τη νέα περίοδο, θα έλεγα με αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Γιατί ούτε στις σχολές, ε, στα σχολεία ε, δεν διδάσκεται στα παιδιά ότι τα πτηνά τρώνε έντομα και αν δεν, τα, αν δεν υπάρχουν έντομα καταστρέφεται η ποικιλότητα. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să o felicit pe colega noastră pentru acest raport și să... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ, Θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο για την έκθεσή της. Όλες οι ιδέες ε, είναι θετικές και τις υποστηρίζω. Ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε να πω, και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Κάποια κράτη-μέλη βλέπουν σαν κάτι αφύσικο τη βιοπικιλότητα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η χώρα μου, η Ρουμανία. Έχει προγράμματα στον τομέα της εξορρυκτικής δραστηριότητας, μεγάλα προγράμματα, μεγάλα έργα Όμως αυτά τα προγράμματα πραγματικά ισοδυναμούν με ένα έγκλημα ε, κατά της βιοποικιλότητας και της φύσης. Σε το σχάρι ένα χρυσορυγείο που πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή Ρώσια Μοντάνα είναι ένα έργο που πραγματικά θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον και οι διαχειριστές αυτοί που θα εκτελέσουν το σχέδιο έδι ξεριζώνουν δέντρα ε, στην περιοχή αυτή. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη πρόληψη και περισσότερο έλεγχο. Αυτό θα πρέπει να κάνει και η Κομισιόν, να μην επιτρέπει να γίνονται καταστροφέ. Είναι κάτι πραγματικά κατεπήγον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και θεωρώ ότι έληξε αυτό το σημείο τη μέησης διάταξη και τώρα μα έχει μείνει και λίγο χρόνο. Γιατί είχαμε προγραμματίσει παρατέταρτο να ξεκινήσουμε τη μήνυα ακρόαση. Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ λοιπόν, μέχρι τις 4 παρατέταρτο. Θα αρχίσει η σύντομη ακρόαση στις 4 παρατέταρτο. Διακόπτουμε λοιπόν από λίγο. Ladies Κυρίες και κύριοι, ξαναρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Είχαμε διακόψει για λίγο, γιατί επρόκειτο να αρχίσουμε την μήνυ ακρόαση με θέμα μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως καθοριστικός παράγων, στις 4 παρατέτατο. Αρμόδιος εισηγητής του Στικάου κυρία Τικάου, συγγνώμη. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τικάου για να ξεκινήσει, εφόσον εκείνη είναι η συγγήτρια για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο, κυρία Τικάου. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες ε, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για την ακρόαση αυτή. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αν θέλουμε να έχουμε μια εσωτερική ψηφιακή αγορά. Και για αυτό το λόγο ανυπομονώ για όλες τις παρεμβάσεις των εμπειρογνωμονών σήμερα, γιατί θέλουμε η έκθεση μας ε, για την ε, ηλεκτρονική κυβέρνηση ως ε, καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαγορά. Θέλουμε ουσιαστικά με την έκθεση αυτή να έχουμε μία εισαγωγή για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να δούμε πώς ε, έχει κατάσταση, ποια είναι τα εμπόδια που έχουν προσδιοριστεί και στο εσωτερικό των ε, κρατών μελών αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί θέλαμε να πετύχουμε, θα θέλαμε να πετύχουμε την ε, διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θέλουμε να εντοπίσουμε τους κυρίους παράγοντες που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για δίκτυα επικοινωνιών, για τα απαραίτητα συστήματα επικοινωνίας, και επίσης θα μιλήσουμε και για συστήματα πληροφορικής που χρειαζόμαστε. Θα συζητήσουμε και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη των διάφορων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες ευρωπαϊκές οδηγίες ισχύουν, και πώς έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Επίσης ε, θα αναφερθούμε στην ηλεκτρονική υπογραφή και στην αμοιβαία αναγνώριση των υπογραφών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μιλήσουμε για την αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και με τις τρίτες χώρες. Θα μιλήσουμε για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας και θα ήθελα να σας πω ότι από το 2001 Είχαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο ό,τι αφορά την εφαρμογή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το 2003 η Κομισιόν παρουσίασε 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται και μέσω ηλεκτρονικών μέσων και οι οκτώ σκόπευαν στο επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 12 στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ορισμένες υπηρεσίες είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικές. Αναφέρομαι στα ηλεκτρονικά συστήματα για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις δημόσιες προμήθειες. Έχουν ε, ωφελήσει τα μάλα κατόπιν της εισαγωγής τους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να πληρώσει κάποιος τους φόρους τους με την, ε, για τις ηλεκτρονικές οδού. Και μπορούμε εδώ να αναφέρουμε και τις ευφύης ε, υπηρεσίες μεταφορών και ακόμη και τα ευφυή e ενεργειακά δίκτυα. Έτσι λοιπόν ε, η εφαρμογή αυτών των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα, έχουμε ιδιαίτερα ευρεία διαδεδομένη εφαρμογή και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για την τροποποίηση του εφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε καλύτερα αυτές τις ε, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, Έχουμε κατά νου και τη δημιουργία μιας νέας υποδομής ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Και εδώ ενυπομονούμε να ακούσουμε, να δούμε την παρουσίαση της πρότασης της Κομισιόν που θα επέλθει του χρόνου και καλύπτουμε και το θέμα των ε, δικτών επιδόσεων. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα αυτό, αλλά και τις χρηματοοικονομικές πόρους και τη διεθνή συνεργασία. Όπως βλέπετε, η έκθεση βασίζεται σε τρεις ανακοινώσεις της Κομισιόν. Η μία αφορά την ε, υιοθέτηση ηλεκτρονικού τιμολογίου ή invoice ε, ως ε, μια εκούσια πρωτοβουλία, αλλά σε επίπεδο ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και την ανακοίνωση για το σχέδιο δράση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ανακοίνωση τη Κομισιόν για το πλαίσιο διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ε, Λόγω σας είπα, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε και την κατάσταση, το state of place, ό,τι αφορά την εφαρμογή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα διάφορα κράτη-μέλη, για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες ε, και ποια μπορεί να είναι τα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Ποια είναι τα εμπόδια στην ε, διαλειτουργικότητα, των υπηρεσιών των διάφορων κρατών μελών και επίσης θα πρέπει να προσδιορίσουμε, να εντοπίσουμε από κοινού αυτούς τους καταλητικούς παράγοντες που θα μπορούσαν ε, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση θα δοθεί προς μετάφραση αρχές Ιανουαρίου. Στις 6 Φεβρουαρίου στην ε, Επιτροπή ΙΤΡΕ θα συζητήσουμε την έκθεση και στη συνέχεια στις 15 Φεβρουαρίου θα έχουμε την καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Νομίζω ότι τα όσα κάνουμε εδώ μέσω αυτής της μήνυα Κρόασης και μέσω της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι φορά... Ε, την ανάπτυξη τη ηλεκτρονικών, ε, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ε, ως καθοριστικού παράγοντα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει τα εμπόδια που βλέπουμε σήμερα και που μα εμποδίζουν να έχουμε υπηρεσίε ηλεκτρονική διακυβέρνηση που να είναι πράγματι διαλειτουργικές και διασυνοριακές. Θα σταματήσω εδώ γιατί θα ήθελα να δώσω το λόγο στου εμπειρογνώμονε. Νομίζω ότι μόνο από κοινού μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτής της φιλόδοξης έκθεσης η οποία πράγματι θα μας ε, δώσει κάποιες σταθερές βάσεις για την ε, μελλοντική ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και κατευθείαν δίνω το λόγο στον κύριο Χουάν Αρέγγι Μακίγιον που είναι υπεύθυνο έργου για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες από τη Γενική Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινωνίας Πληροφορίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την δυνατότητα να είμαι εδώ σήμερα στη μήνυ αυτή ακρόαση. Να ευχαριστώ και την κυρία Τσικάου. Άκουσα τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, κυρία Τσικάου, και πραγματικά αυτά που είπατε βρίσκουν σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ό,τι αφορά δηλαδή συνολικά τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και ειδικότερα της ανάπτυξης της νέας ψηφιακή αγοράς. Είχα προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες, τις οποίες φαντάζομαι ότι θα βλέπετε σύντομα στην οθόνη. Όπως είπα, χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ελπίζω με την παρουσίασή μου να σας δώσω μια καλή εικόνα της κατάστασης που θα σας βοηθήσει να εκπονήσετε και την γνωμοδότησή σας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Εγώ θα σας μιλήσω για το σχέδιο δράσης ηλεκτρονική διακυβέρνηση το οποίο εγκρίθηκε προενός έτους. πρώτη επέτειο του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Ένα χρόνο έκλεισε το σχέδιο αυτό. Για να δούμε, θα δούμε και τις διαφάνειες κάποια στιγμή. Uh, uh, να, ένα επιχείρημα να υπάρξει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν τώρα και τις διαφάνειες. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο δράσης. Είχαμε ένα από το 2006 στο 2010. Όλα τα κράτη-μέλη σημείωσαν σταθερή πρόοδο για την υλοποίηση της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τις επιγραμμικές υπηρεσίες, και ούτω καθεξής. Άρα, η ερώτηση είναι, χρειαζόμαστε ένα ακόμη πρόγραμμα. Είδαμε ότι παρέμεναν κάποιες σημαντικές προκλήσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις στον αριθμό. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και ανάγκη για άνοιγμα και διαφάνεια από πλευράς ε, των διοικήσεων. Ένα πολύ ισχυρό αίτημα επίσης, ε, το οποίο ε, διατυπώνεται από τις επιχειρήσει από του πολίτε να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητε, ε, το λεγόμενο empowering, ενδυνάμωση. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης. Τρίτη προτεραιότητα, πολύ σημαντική θα πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά, την ψηφιακή ενιαία αγορά. Τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν αντιλαμβάνονται ότι με την ε, ανάπτυξη λύσεων και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επειδή δεν υπήρξε συνεργασία, τελικά αυτό που έγινε ήταν ότι ορθώθηκαν φραγμοί εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν δηλαδή κάποιοι υλικοί φραγμοί και δημιουργήθηκαν ψηφιακοί φραγμοί και πρέπει να μην δρούμε απομονωμένο ένας από τον άλλο, γι' αυτό αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ψηδέ και του χρηματοοικονομικού κλίματος είναι προς όφελός μας και μόνο να φροντίσουμε να είναι ο δημόσιος τομέας βιώσιμος αποτελεσματικός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική όθηση που στηρίζει την εξέλιξη αυτή. Όπως είπα, από τη δική μας πλευρά η συγκεκριμένη μεταφορά στην δράση είναι η δρομολόγηση του σχεδίου δράσης πέρυσι, τέτοια εποχή και αυτό το σχέδιο δράσης ήταν αποτέλεσμα μιας υπουργικής διάσκεψης ε, στο Μάλμο το 2009. Όλοι οι Υπουργοί όλων των κρατών μελών στήριξαν και εξέφρασαν την πολιτική τους δέσμευση προς ένα νέο σχέδιο δράσης για την λιτωνική διακυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό στήριξε και ένας πολύ σημαντικός παίκτη, η βιομηχανία. Και για πρώτη φορά υπήρξε και δήλωση των πολιτών Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, οι πολίτες τόνισαν ε, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τέσσερις ήταν οι πολιτικές προτεραιότητες. Η ενδυνάμωση των χρηστών, ενίσχυση της ενίας αγοράς, ώστε να τον πιο αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τέλος η ανάπτυξη των προϋποθέσεων για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα τα προηγούμενα. Δηλαδή ηλεκτρονική ταυτότητα, ηλεκτρονική υπογραφή, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, δηλαδή αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στο χρήστη, το λεγόμενο cloud computing και ούτω καθεξής. Ώστε αυτό το όραμα του Μάλμε να γίνει πραγματικότητα, να πάρει σάρκα και οστά. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια τη σχέση, τη διασύνδεση μεταξύ της δήλωσης του Μάλμε και της ψηφιακή, του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης λοιπόν έχει δύο κυρίους, αν μου επιτρέπετε, τους οποίους υπηρετεί. Έχετε λοιπόν εδώ τις τέσσερις προτεραιότητες με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Για την πρώτη προτεραιότητα λοιπόν, τι εννοούμε να δώσουμε περισσότερη δύναμη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εννοούμε να έχουμε χριστοκεντρικές υπηρεσίες, το χρήμα ΙΤΑ, να έχουμε παραγωγή συνεργατική. Δεν ξέρω αν βλέπετε καλύτερα, γιατί εγώ δεν βλέπω τόσο καλά. Είναι λίγο μικρά τα γράμματα. Λοιπόν, ε, συνεργατική παραγωγή υπηρεσιών, δηλαδή να ανοίξουμε πόρτες παράθυρα της ε, διακυβέρνησης και της δίκησης ε, σε τρίτους που να μπορούν και αυτοί να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να παράγουν υπηρεσίες οικονομικής διακυβέρνησης κοινοτοπολιτών, ιδιώτες. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ταλέντο και πολλή γνώση εκεί έξω και η διοίκηση, ε, η κεντρική, πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται τι δυναμικό υπάρχει. Άρα με τη συνεργασία με τρίτους και με την κοινωνία των πολιτών μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερες υπηρεσίε για όλους. Η επανάχρηση πληροφοριών στον δημόσιο τομέα πολύ σημαντικό σκέλος αν θέλουμε να έχουμε πιο διαφανή ανοιχτή διακυβέρνηση, αλλά δημιουργούμε και επιχειρηματικές ευκαιρίες για να μπορέσουν οι προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν ε, τη μεγάλη μάζα πληροφοριών που, έχει, υπάρχουν στο επίπεδο της δίκησης για να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και νέες εφαρμογές. Μεγαλύτερη διαφάνεια και όλα αυτά θα διευκολύνουν και τη συμμετοχή των πολιτών στην χάραξη πολιτικής, στις νομοθετικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Όλοι δηλαδή εντάσσονται καλύτερα και περισσότερο σε αυτές τις διαδικασίες. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Σας μίλησα πριν για κάποια εμπόδια, για τους φραγμούς που ορθώθηκαν αλλά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στόχο έχει να κάνει πιο εύκολη την ζωή μας. Δηλαδή με λίγα πατήματα κουμπιών να μπορούμε να φέρουμε σε πέρας κάποιες διαδικασίες. Στα κράτη-μέλη αυτό μπορεί να ισχύει εντός των κρατών μελών δηλαδή. Αλλά αν θέλουμε αυτό να το κάνουμε και σε άλλες χώρες, είτε αυτό δεν γίνεται δυνατόν, είτε καθίσταται πολύ δύσκολο γιατί πρέπει κανείς να παρίσταται, να πάει αυτοπροσώπως κάπου ή να στείλει κάποια χαρτιά κτλ. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ε, πάρα πολύ απρόσκοπτες ε, υπηρεσίες, ε, προσωπική κινητικότητα, να μπορούν δηλαδή πολίτες να μετακινούνται ανά την Ευρώπη πιο εύκολα από ό,τι μέχρι τώρα, να μπορούν δηλαδή να διαμένουν κάπου, να εγκατασταθούν, να ε, είτε για να εργαστούν είτε για μετά τη σύνταξή τους, οπουδήποτε. Και να μην έχουν πρόβλημα με τις υπηρεσίες να μπορούν ηλεκτρονικά όπως και στη χώρα τους να δεκπεραιώνουν κάποιες διαδικασίες. Και τέλος, τρίτο σημείο, διασυνοριακές υπηρεσίες. Ένας από τους στόχους του σχεδίου δράσης είναι μέχρι το 2015 να έχουμε διασυνοριακές υπηρεσίες διαθέσιμες online. Τρίτο στόχο είναι η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα. Αυτό τι θα πει. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι τεχνολογίες των επικοινωνιών και των πληροφοριών αλλάζουν τις διαδικασίες τις οργανωτικές. Δεν είναι απλά δηλαδή να έχουμε κάποια στοσελίδα στη διάθεσή μας ε, και να ανεβάζουμε, να αναρτούμε εκεί κάποια έντυπα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να υπάρχει πραγματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θέλουμε λοιπόν να ξανασκεφτούμε και να αναδιορθώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Φυσικά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να φαίνεται ότι μειώνει και το διοικητικό άχθο. Πρέπει να συμβάλλει σε αυτό, είναι ε, σαφές. Επίσης, έχει και τις δυνατότητες ε, να κάνει πιο πράσινη την κυβέρνηση τη διακυβέρνηση μάλλον, δηλαδή ε, να είναι μειωμένα ο χρόνος μετακίνησης και ούτω καθεξής, ε, να μην υπάρχουν ε, τόσα χαρτιά. Και ένα τελευταίο στοιχείο που στηρίζει και όλα τα προηγούμενα είναι οι προϋποθέσεις. Δηλαδή προδιαγραφές, διαλειτουργικότητα, πάρα πολύ σημαντική. Οι βασικοί παράγοντες, οι enablers, ηλεκτρονικές ταυτότητες, υπογραφές όπως είπα και τέλος η καινοτόμος ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα αξιοποιεί το δυνατόν, που θα αξιοποιεί δυνατόν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Τι μέσα λοιπόν έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα για την Κομισιόν ε, κατά την νομοθετική έννοια, αλλά από το 2000 και μετά τα κρατη συμφώνησαν ότι είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι προ όφελο όλων των κρατών μελών να συνεργάζονται προ την επίτευξη ορισμένων κοινών στόχων. Έχουμε λοιπόν τα μέσα πολιτική με αυτό το σχέδιο δράση, υπουργικέ διασκέψει επίση με τη στήριξη λοιπόν από το υψηλό επίπεδο και πριν από ένα μήνα είχαμε την έκτη Υπουργική Διάσκεψη στο Πόσναν και κάτι πολύ σημαντικό είναι και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η συγκριτική αξιολόγηση, benchmark, να δούμε δηλαδή πού βρισκόμαστε, ποια πρόοδο έχει επιτευχθεί και ούτω καθεξής. Και χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία χρειάζονται. Ε, πρώτα απ' όλα έχουμε την έρευνα, έχουμε τα διάφορα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα, με τελευταίο το έβδομο όπου εκεί υπήρχε στόχος ε, τεχνολογίες πληροφοριών επικοινωνιών για τη διακυβέρνηση και την μοντελοποίηση πολιτικής και η ανάπτυξη με τα διάφορα προγράμματα στήριξης πολιτικής στον τομέα πάντα των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα για να δείτε τις προτεραιότητές μας. Μία από αυτές είναι λοιπόν η ενίσχυση της ε, εσωτερικής αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε σε απρόσκοπτε υπηρεσίε ε, διασυνοριακά, θέλουμε να υπάρχει ένα κοινό κατάλογο βασικών διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών και θέλουμε να είναι πλήρως διαλειτουργικέ υπηρεσίε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μια τελευταία διαφάνεια και θα έχω ε, ολοκληρώσει εγώ την παρουσίασή μου. Βλέπετε εδώ δύο βασικές δράσεις που θέλω να τονίσω για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, το EID, δηλαδή ηλεκτρονική ταυτότητα και το e-signature, ηλεκτρονική υπογραφή. Σημαντικό στόχο είναι αναθεώρηση τη οδηγία για την ε, ηλεκτρονική υπογραφή. Πρόκειται για τη βασική δράση 3 και έχουμε και τη βασική δράση 16. Θα έχουμε λοιπόν απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση τη ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Θα έχουμε νέα μελλοντικά λοιπόν σε αυτά τα μέτωπα. Αυτή ήταν η δική μου λοιπόν παρουσίαση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Πήραμε τώρα την ενημέρωση από την Επιτροπή και τώρα αν έχετε ερωτήσεις, έχετε την ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Διαφορετικά μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Αν έχετε ερωτήσεις, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. So, I have three short remarks and three questions. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρει σύντομε παρατηρήσει και τρει ερωτήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην προώθηση τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση από το 2005 με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και υπάρχουν και πολλέ μελέτε που ασχολούνται με την διαθεσιμότητα και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη αλλά σε πολλές μελέτες ε, δεν φαίνεται να είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα σε πολλά κράτη-μέλη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπους που δεν καταπολεμούν τη γραφειοκρατία. Πολλά προγράμματα βασίστηκαν στις ίδιες γραφειοκρατικές αρχές Χρησιμοποιούμε μη αποτελεσματικά λοιπόν τη σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργήσουμε επιπλέον γραφειοκρατία και πολλές μελέτες δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα των, ε, ε, τεχνολογιών αυτών έχουν σχέση με την ε, χρήση υπολογιστών και διαδικτύου. Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες χρήσιμο περιεχόμενο για την καθημερινή του ζωή, διαφορετικά δεν θα έχει περιεχόμενο το θέμα της αναθεώρησης της ψηφιακής ατζέντα. Η ερώτησή μου είναι αν έχουν γίνει πρόοδοι για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεύτερον, πώς αξιολογείται τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη-μέλη. Ε, και δεύτερον, τι ε, σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή για να ε, αλλάξει την προσέγγιση της και να δημιουργήσει μια πραγματικά ψηφιακή αγορά ε, υπηρεσιών και τρίτον ποιοι είναι οι μετρήσιμοι στόχοι που έχουν επιτευχθεί για την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τι μετρήσιμους στόχους για το μέλλον έχουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Τικάου. Ε, eu aș vrea să întreb Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Αρεγκή τι οικονομικοί πόροι υπάρχουν για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 για την υλοποίηση των ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης. Δεν αναφέρομαι ε, μόνο στην υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Περισσότερο μιλώ για τη διασφάλιση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας. Υπάρχει το πρόγραμμα για τον ορίζοντα του 2020, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλες γραμμές στα μελλοντικά δημοσιονομικά πολιτικά δημοσιονομικά προγράμματα για αυτές τις υπηρεσίες. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε από αυτό θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαδουρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την εξήγηση. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα κάπως καθυστερημένη και δεν ξέρω αν αυτό που θα ρωτήσω το σχολίασε ο μιλητής ε, στην αρχή της ομιλίας του. Μας υπενθύμησε τις τέσσερις προτεραιότητες που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης ε, και απαιτείται ο καλός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Γίνεται αυτός ο συντονισμός και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Για τον κύριο Τσουκαλά. Να σας πω τώρα ότι οι μετρήσιμοι στόχοι για την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το προηγούμενο σχεδίο δράσης είχε θέσει πολύ συγκεκριμένους στόχους για τις ε, ηλεκτρονικές ε, δημόσιες συμβάσεις ε, και είχαμε πει ότι μέχρι το 2010 100% όλων των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να διατίθενται online και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από το 50% των εταιριών πολύ αισιόδοξο τελικά ήταν, πολύ αισιόδοξο ήταν αυτός ο στόχος. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι ότι η διαθεσιμότητα των ε, ηλεκτρονικών ε, προμηθειών ήταν κάτω από το 60% και δεν ε, έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για το πόσο τελικά τέθηκε σε εφαρμογή ε, αυτή, αυτές τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και επίσης στο σχέδιο δράσης ε, τώρα έχουμε κάποιους πιο ρεαλιστικούς στόχους αν και φιλόδοξοι Μέχρι το 2015, 50% των Ευρωπαίων πολιτών θα έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάποια στιγμή. Και τα στοιχεία που έχουμε από το 2010 είναι ότι περίπου 42% των πολιτών χρησιμοποιούν ε, την υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τα τελευταία χρόνια ήταν ε, πολύ αργή η πρόοδος, αλλά είδαμε ότι το 2010 είχαμε μια σημαντική αύξηση. Ελπίζουμε λοιπόν να συνεχίσει αυτή η τάση και μέχρι το 2015 να έχουμε ξεπεράσει το 50%. Και έχουμε και τον ίδιο δείκτη για τις επιχειρήσεις. 80% ε, των επιχειρήσεων έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τώρα είμαστε περίπου στο 60%. Έτσι λοιπόν, ε, ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε και το στόχο αυτό. Τώρα, πώς ε, μετράμε τη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όπως ε, είπε και η κυρία Τικάου, αναφέρθηκε στις 20 ε, δασικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες επιγραμμικά. Από το 2001 γίνονται μετρήσεις για το θέμα αυτό και βλέπουμε τώρα ότι χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε τότε, οι στόχοι ήταν ε, γενικά επιτυχής. Ε, αυξηνόμενος, ε, αυξήθηκε ο αριθμός των χωρών όπου είχαμε διαθεσιμότητα αυτοϋπηρεσιών και φτάναμε είτε στο 100%, σχεδόν στο 100% είτε στο 100%. Φυσικά υπήρχαν κάποιες αποκλήσεις μεταξύ των χωρών. Αλλά η τάση είναι ότι όλες οι χώρες σημειώνουν σταθερή πρόοδο στη χρήση των δικτών αυτών. Ως προς ε, τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρησιμοποιούμε τις ε, μελέτες της Eurostat. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία της Eurostat με τα στοιχεία των εθνικών Συνδρυμάτων ε, συλλογή στατιστικών στοιχείων με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Τώρα για την ερώτηση για τους δημοσιονομικούς σπόρους που θα έχουμε για την περίοδο 2014-2020 η Κομισιόν πρότεινε ως ε, τμήμα του ορίζοντα 2020 του, το Connecting Europe Facility, δηλαδή έχουμε αυτό το μέσο το οποίο στοχεύει στο να αναπτύξει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, επικοινωνιών και ICT ε, τις τεχνολογίες ε, επικοινωνιών και πληροφοριών και κυρίως αναφέρομαι στις ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και το κονδύλι για το τμήμα τεχνολογιών ε, και επικοινωνών και περιφερειών είναι 9,2 δισεκατομμύρια περίπου και από αυτά η Κομισιόν προτείνει από αυτά τα 9,2 να έχουμε 2 δις για την ανάπτυξη των διασυνοριακών ε, υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως ε, σε τομείς όπως ε, οι ηλεκτρονικές δημοσίες προμήθειες, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτλ. Η πρόταση της Κομισιόν εστάλει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θα συζητηθεί τώρα και στα υπόλοιπα όργανα. Και για την κυρία Μαδουρέλ. συντονισμός με τα κράτη-μέλη. Είναι αλήθεια, θα έπρεπε να το έχω αναφέρει ως πέμπτη προτεραιότητα ίσως του σχεδίου δράσης. Βεβαίως έχει το δικό του κεφάλαιο στο σχέδιο δράση ε, υπό του όρου τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αν δεν συνεργαστούν τα κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια Υπήρχε προθυμία συνεργασίας. Στην προηγούμενη στρατηγική είχαμε την υπομάδα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τώρα ω τμήμα του ψηφιακού θεματολογίου έχουμε το e-government group, αυτή την ομάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών και αναλύουν ε, την ε, πρόοδο, ανταλλάσσουν εμπειρίες ε, και εξετάζουν αν ο ρυθμός της, ε, της πρόοδου είναι επαρκής ή αν οι πολιτικές ε, προτεραιότητες που είχαν τεθεί στο παρελθόν ξεκολουθούν να ισχύουν κτλ. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, είναι σημαντικοί πρωταγωνιστές και ο συντονισμό είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες του σχεδίου δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ομιλιών και ερωτήσεων και θα ήθελα να λάβουν θέση τώρα ο κύριος Κατινά, ο κύριος Μισελ Κατινά και ο κύριος ε, Πίτερ Μπάινε Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο γύρο. Ξεκινάμε λοιπόν με το δεύτερο θέμα που είναι το πώς θα τλήσουμε τα ωφέλη από την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε τον κύριο Μισελ Κατινά και τον κύριο Πίτερ Μπράινε. Έχουν 10 λεπτά ο καθένας για να μας αναπτύξουν τις θέσεις τους και μετά θα υποβάλουμε ερωτήσεις. Κύριε Κατινά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τικάου. Εκπροσωπώ δύο γενικέ διευθύνσει που είναι υπεύθυνε για το θέμα τη ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εκπροσωπώ τη δική μου Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανία, αλλά και την Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσιών. Το πρώτο μου μήνυμα λοιπόν θα είναι το ότι θέλω να επιμείνω ε, για το πόσο συνεισφέρει αυτή η πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία διαρθρωτική που στόχος της είναι να οδηγήσει τις επιχειρήσεις να θεσπίσουν ολοκληρωμένα και ψηφιακά συστήματα για όλες τους τις συναλλαγές. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι μια θεμελιώδης προσπάθεια για τις επιχειρήσεις. Ε, βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων κάθε επιχειρήσεως, μικρής ή μεγάλης και συνδέεται, συνδέει τα παραγωγικά του συστήματα και τα χρηματοοικονομικά του συστήματα καθώς και τα λογιστήριά τους. Περνάμε λοιπόν στο ψηφιακό κόσμο με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Με αυτό το πέρασμα στον ψηφιακό κόσμο θα μπορέσουμε να δρέψουμε και τα ωφέλη και την αποτελεσματικότητα. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα δίνουν τη δυνατότητα σε πιο σύντομο διάστημα πληρωμών, σε μικρότερους κινδύνους, σε μείωση του κόστους διεκπαιρέωσης και θα υπάρχει ε, το πέρασμα στην ψηφιακή, στην πλήρως ψηφιακή εποχή. Θεωρούμε σήμερα ότι μόνο 10% του συνολικού όγκου τιμολογίων που ανταλλάσσονται μεταξύ επιχειρήσεων γίνονται με ολοκληρωμένο ψηφιακό τρόπο. Οι δυνατότητε τη ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μεγάλε, αλλά δεν τι έχουμε εκμεταλλευτεί αρκετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικοί φραγμοί και χρειάζεται τυποποίηση. Υπάρχουν ε, και ρυθμιστικοί φραγμοί που επίσης περιορίζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι, το Δεκέμβριο του 2010, ενέκρινε μια ανακοίνωση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση με ένα πρόγραμμα δράσης, ώστε η ηλεκτρονική τιμολόγηση να γίνει ο κύριος τρόπος τιμολόγησης στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Αυτό το σχέδιο δράσης έχει τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο που δεν θα έχει διακριτική μεταχείριση για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Και όπως γνωρίζετε το τωρινό πλαίσιο ε, ε, είναι εις βάρος της ε, ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δεύτερος πυλώνας θα είναι να υποστηρίξουμε τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ξέρουμε ότι αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει το χρησιμοποιήσουν, θα μπορέσουμε να πούμε ότι οι περισσότερε επιχειρήσει θα έχουν πλέον κινηθεί προ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Τρίτο πυλώνας, να δημιουργηθεί ένα διαλειτουργικό περιβάλλον. Επανερχόμαστε σε αυτό το μόνιμο στη μόνιμο εποδό της διαλειτουργικότητας. Και τέταρτος πυλώνας, να έχουμε κοινά πρότυπα, να προωθήσουμε την έγκριση κοινών προτύπων. Εδώ και ένα χρόνο οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν δουλεύουν προσπαθώντας να να υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις. Έχουμε σημαντικές πρόοδους κατά τη γνώμη μου και από νομικής πλευράς, διότι εδώ έχει εγκριθεί η νέα οδηγία για το ΦΠΑ που εγκρίθηκε το 2010, που κατήργησε τη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των τιμολογίων σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει επεξηγηματικά δελτία για να διευκολύνει την κατανόηση των νομικών κειμένων και για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή μεταφορά της οδηγίας από τα κράτη-μέλη σε εθνική νομοθεσία. Όσον αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή, ξέρετε ότι η φυστάμενη οδηγία δημιουργεί προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί ότι θα αναθεωρήσει την οδηγία αυτή ξεκινώντας από το 2012. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα, την έγκριση του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τομεακά προγράμματα με πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Αυτά τα προγράμματα συνίσταται στο να δημιουργηθεί μαζί με τη βοήθεια των παρόχων υπηρεσιών να δημιουργηθούν πλατφόρμες πληροφόρησης μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή ανατομέα θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών θα αμείβονται για να δημιουργούνται αυτές οι πλατφόρμες διαλειτουργικότητας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διατηρούν το, το ψηφιακό τους σύστημα και θα δημιουργείται το κατάλληλο σύστημα διεπαφής, interface, με τους ε, προμηθευτές ε, ε, ή εντολής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα, διευκολυνθούν, θα διευκολυνθεί η δημιουργία αυτών των ηλεκτρονικών πλατφορμών τέτοιες πλατφόρμες διαλειτουργικότητας έχουμε δει στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των logistics και των μεταφορών και το 2012 θα έχουμε στον τομέα του τουρισμού και της βιομηχανίας τροφίμων. Όσον αφορά τους πυλώνες 3 και 4, θα είμαι σύντομος γιατί ο Πίτερ Μπράιν θα αναφερθεί λεπτομερέστερα. Αφορούν αυτοί οι πυλώνες την τυποποίηση και εδώ θέλουμε να ζητήσουμε από τους οργανισμούς τυποποίησης πρώτον να διευκρινίσουν τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά τους ελεγκτές ή όσον αφορά την τήρηση φορολογικού δικαίου και σε αυτούς τους πυλώνες, τον 3 και τον 4, θα ζητήσουμε από τους οργανισμούς τυποποίησης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης να ακολουθήσουν μια σύγκληση σημασιολογική. Δηλαδή όταν θα υπάρχει ανταλλαγή ηλεκτρονικού τιμολογίου να υπάρχει τυποποίηση των στοιχείων που θα περιλαμβάνονται σε ένα τιμολόγιο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι πληροφορίες πρέπει να δίνει μια επιχείρηση στο τιμολόγιο της. Πρέπει οι πληροφορίες αυτές να είναι τυποποιημένες, να είναι οι ίδιες. Και όσον αφορά την τεχνολογική διαλειτουργικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο εύκολη, διότι έχουμε πολύπλοκα ψηφιακά συστήματα που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα. όμως τα αντελασσόμενα δεδομένα θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, γιατί δεν μπορούμε ε, να να έχουμε διαφορετικά στοιχεία. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε τη διεύθυνση, παραδείγματο χάρη, και την επωνυμία μια επιχείρηση. Αυτά είναι βασικά δεδομένα. Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να δεσμευθούν υπέρ τη ηλεκτρονική. Ε, τιμολόγησης και στα κράτη-μέλη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν εθνικά φόρουμ για την ε, ψηφιακή τιμολόγηση και αυτά τα φόρουμ θα υποστηρίζουν ε, την εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου σε εθνικό επίπεδο θα συμμετέχουν οι βασικοί φορείς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα εντοπιστούν τα προβλήματα, θα υποβληθούν προτάσεις ε, και θα προταθούν λύσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. 18 κράτη-μέλη έχουν φόρουμ. Η Ιταλία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Η Ιταλία νομίζω αυτή τη στιγμή τα ολοκληρώνει και η Γαλλία πολύ σύντομα. Επομένως 20 κράτη-μέλη θα έχουν ολοκληρώσει τα εθνικά φόρουμ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση όπου συνενώνονται οι εκπρόσωποι των εθνικών φόρουμ και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς που θεωρούνται δασικοί ε, και αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ θα ανταλλάσσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πληροφορίες και θα κάνει μια διάγνωση της κατάστασης και θα λάβει και τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεράσουμε τα κυριότερα εμπόδια προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το Σεπτέμβριο του 2011 έγινε μια πρώτη συνεδρίαση αυτού του φόρουμ στις Βρυξέλλες ε, και δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες εργασίας που μέχρι το καλοκαίρι του 2012 θα υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή και θα συζητήσουμε μέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ αυτές τις προτάσεις και η Επιτροπή με βάση αυτές τις συστάσεις θα συνεχίσει με σκοπό την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων για την θέσπιση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Θέλω να τονίσω τη σημασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ιδίως στο πλαίσιο Τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δέσμευση ότι θα προωθήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνη τη. Χρειάζεται υποστήριξη και από τα κράτη-μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο έτσι θα μπορέσει η ευρωπαϊκή τιμολόγηση να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπράινε. Uh, good afternoon everyone. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Τικάμου για την πρόσκληση. Και εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ που άκουσα τόσα είπε ο κύριο Κάτινα γιατί συναντηπλήρωσε με τη δική μου άποψη. Λέγομαι Πιτεμπράν, είμαι η διευθυντή τη PricewaterhouseCoopers ε, και ε, επίση είμαι επικεφαλή ε, του δικτύου Archive και Επίσης, έχω βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της, ε, των προγραμμάτων ε, των σχετικών project για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Να δούμε την ε, πρώτη διαφάνεια. Στο πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει δυνατότητα για εξοικονόμηση σε περίοδο εξιετών 243 εκατομμυρίων ευρώ και στο Βέλγιο υπολογίσαμε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε λοιπόν πολλές μελέτες και είναι τεράστια τα ποσά που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, αλλά κατόπιν βλέπουμε ότι η συνολική οθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγηση σε όλη την Ευρώπη είναι κάτω του 15%. Είναι κάπως περίεργο λοιπόν. Αν και έχουμε όλη αυτή τη δυνατότητα εξοικονόμησης, έχουμε λιγότερο από 15%. Υπάρχει τεχνολογία και η νομοθεσία το επιτρέπει. Και αυτό που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα προβλήματα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια θέση είδου ε, κάτσε 22 Δηλαδή, οι δικοί μου προμηθευτές δεν μπορούν να στείλουν ε, ηλεκτρονικά ε, τιμολόγια, ούτε οι πελάτες που δεν μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Και έτσι λοιπόν εγώ δεν συμμετέχω και θα έλεγα ότι αυτό δημιουργεί κάποια εμπλοκή, γιατί τελικά ποτέ δεν προχωρούμε ενώ λοιπόν δεν θα συμμετάσχω. Βασικά λοιπόν ε, αυτός ο όγκος θα πρέπει να αυξηθεί ε, έτσι ώστε να έχουμε πραγματική ηλεκτρονική τιμολόγηση και θα πρέπει να έχουμε τρία τεινά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ανοιχτά πρότυπα και να προωθήσουμε τη χρήση των ανοιχτών προτύπων. Ε, νομικές απαιτήσει πρέπει να απλουστευτούν. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, η διαδικασία απλουστευσης έχει ήδη ξεκινήσει. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι επίσης ε, οι κυβερνήσεις ε, να δίνουν ε, το ηγετικό παράδειγμα. Τώρα, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια για τη χρήση των ανοιχτών προτύπων. Εδώ πρέπει να επιλύσουμε αυτό που αποκαλώ εγώ το παράδοξο της τυποποίησης. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Παράδοξο τυποποίησης λοιπόν, έχουμε τόσο πολλά πρότυπα και τελικά δεν έχουμε κανένα. Έχουμε λοιπόν το GCS Fact, έχουμε το ISO 22 ε, για τον ε, χρηματοοικονομικό τομέα και ξέρουμε ότι γίνεται και πολλή δουλειά έτσι ώστε να υπάρχει σύγκληση αυτών των προτύπων αλλά όλη αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Και θα έλεγα ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και όλοι όσοι μπορούν θα έπρεπε να προσπαθήσουν ε, να δώσουν μια όθηση σε αυτή τη διαδικασία σύγκλησης έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα και μόνο καθολικό πρότυπο. Όταν ε, μιλάμε τώρα για τις νομικές απαιτήσει, ε, μιλάμε για τις απαιτήσει ΦΠΑ, για την έκδοση τιμολογίου. Έτσι λοιπόν, βάσει της μελέτες που υλοποιήσουμε για την ΓΑΜΑ για το 2008, το 2008 μάλλον, όταν εισαγάγαμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης ε, μεταξύ των ε, τιμολογίων, των ηλεκτρονικών και των τιμολογίων σε χαρτί και αυτό σημαίνει βασικά ότι τεχνολογικές απαιτήσει ε, αφαιρέθηκαν από την προηγούμενη οδηγία και αυτό σημαίνει ότι ο υποκείμενο στο φόρο είναι αυτό που θα καθορίσει την αυθεντικότητα και την ακαιρεότητα. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό για τι επιχειρήσει, ότι δηλαδή είναι ελεύθερο κάποιο ε, να επιλέξει με ποιο τρόπο θα κάνει τη ε, τις δικές του επιχειρήσεις ε, και να διαλέξει πώς ποια διαδικασία θα ακολουθήσει και να υποφεληθεί πλήρως. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 2010 με τη δημοσίευση της οδηγίας, αλλά θα πρέπει να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Θέλω να ζητήσω λοιπόν από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο ε, να διασφαλίσουν ότι τα κράτη-μέλη στις εθνικές νομοθεσίες ε, θα μεταφέρουν πλήρως την οδηγία θα σεβαστούν το πνεύμα της οδηγίας, δηλαδή σε μεταχείριση και να μην υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσει, καμία πρόσθετη απαίτηση. Και περνάμε και στο τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό. Οι κυβερνήσει ε, που θα δίνουν ε, το καλό παράδειγμα. Εδώ οι κυβερνήσει έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και εγώ Συμμετέχω στο project ε, η prior που ξεκίνησε το 2007 από τη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν για την Πληροφορική, το e-prior. Είναι μια υποδομή που επιτρέπει τους προμηθευτές ε, να στείλουν τιμολόγια ηλεκτρονικά προς την Κομισιόν ε, με έναν ε, εντελώς ολοκληρωμένο τρόπο και παράλληλα έχουμε το Project PEPOL το οποίο επιτρέπει σε οποιαδήποτε δίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε ηλεκτρονική σύναψη δημοσίων συμβάσεων και στην έκδοση ηλεκτρονικών τελογίων και το υπέρ έχει συνδεθεί με την υποδομή PEPOL και αυτό είναι ένα πολύ καρό παράδειγμα της διαλειτουργικότητας ε, των ε, δύο κυρίων αυτών ε, project για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, αυτή η λύση είναι μια λύση που βασίζεται στο δίκτυο, είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στο δίκτυο. Οι εταιρείε μπορούν να στείλουν τιμολόγηση XML, τιμολόγια XML, αλλά και για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι μια λύση εύχριστη Έχουμε λοιπόν αυτή την πύλη για τους προμηθευτές. Μία μικρή εταιρεία μπορεί να ε, κάνει λογκόν, ε, να μπει στο σύστημα για να στείλει ηλεκτρονικά τιμολόγια πολύ εύκολο, με πολύ εύκολο τρόπο. Και σε ό,τι αφορά το rollout, την ανάπτυξη, 30 προμηθευτές έχουν συνδεθεί τώρα ή θα είναι συνδεδεμένοι με το e-prior Σύντομα, αυτό που βλέπουμε ε, στην πράξη είναι ότι καθυστερεί κάπως η διαδικασία, είναι κάπως αργή. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στις συμβάσεις μια ρήτρα που επιτρέπει στην Κομισιόν να υποχρεώσει αυτούς τους προμηθευτές να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και αυτό το έκανε η Κομισιόν. Και η ε, τώρα υποχρεώνει τους προμηθευτές να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και εδώ βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε και παρόχους ε, υπηρεσιών, service providers. Ε, ζητείτε από τους προμηθευτές να στείλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προς αυτό το σύστημα e-prior, αλλά πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν κάποιο πάροχο υπηρεσία και η Κομισιόν πρέπει να συνεργάζεται με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών έτσι ώστε να ε, έχουμε ωφέλη και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και κάτι τελευταίο που το βλέπετε κάτω-κάτω, σήμερα έχουμε την Digit και την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Πασχόλησης που χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα. Και θα ήθελα να προτείνω την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση του πράιρου στο ιστορικό της Κομισιόν, έτσι ώστε όλες ε, οι δέλτα και όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι υπηρεσίες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ε, τις ηλεκτρονικές προμήθειες έναντι των προμηθευτών τους. Να σας πω ότι είμαι και μέλος ε, του Βελγικού Φόρουμ για την Ελεκτρονική τιμολόγηση που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ε, Φόρουμ που, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κατινάκ και μπορώ να σας πω ότι το Βελγικό Φόρουμ βλέπει, παρακολουθεί ανυπόμονα το τι σημαίνει στην Ευρώπη ε, και προσπαθούμε φυσικά να μάθουμε όσο δυνατόν περισσότερα από τα ευρωπαϊκά όργανα, του ευρωπαϊκού θεσμού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο Κομισιόν να συνεχίσουν να δίνουν ε, το καλό παράδειγμα προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ακριβέστερες πληροφορίες που μας δώσατε και δίνω το λόγο στους ομιλητές για ερωτήσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς. Είστε ο πρώτος ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και νομίζω ότι οι δύο ομιλητέ του θέλω να ευχαριστήσω, ουσιαστικά με κάλυψαν. Θα αναφέρω πάντως δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση τι πρέπει να γίνει ώστε η ηλεκτρονική τιμολόγηση να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιος είναι ο ρόλος των κοινών τεχνικών προτύπων σε όλη αυτή την ιδέα. Η κυρία Χέρτσογκ. Όχι, συγγνώμη, κυρία Τικάου. Συγγνώμη, λάθος μου λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι ε, ο κύριος Κέλλη θα θέλει και αυτό το λόγο. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση. Από το 2009 και μετά, εξ όσων γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στους ε, ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ε, να καταλήξουν σε ένα κοινό πρότυπο για τα τιμολόγια. Θυμάμαι ότι είχαμε τις ακροάσεις του Επιτρόπου Ταγιάννη και του είχα θέσει ερώτημα τότε για την ε, πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την πρόθεση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είναι πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να περιμένουμε το σχέδιο δράσης που θα επιταχύνει την εισαγωγή και καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν όλα τα συστήματα δημοσίων προμηθειών να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Και στο Μάντσεστερ είπαμε ότι μέχρι το 2015 το 15% των ηλεκτρονικών προμηθειών να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα συστήματα δημόσιων προμηθειών να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν και ένα καλό παράδειγμα να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις και φαντάζομαι ότι τις χώρες θα τις ενδιαφέρει να ακολουθήσουν το σύστημα αυτό της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη αλληλεπίδραση ε, και σχέση με την αγορά των δημοσίων προμηθειών. Έχουμε δει μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δείχνουν ότι για κάθε τιμολόγιο εξοικονομούνται 6 ευρώ. και μειωμένη ε, είναι η ρήπανση, λιγότερο το χαρτί που χρησιμοποιείται. Οι δε αρχές επίσης ε, κάνουν κάποιες οικονομίες, είναι λιγότερα τα σφάλματα, όλα αυτά τα ωφέλη, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν και ένα οικονομικό και ένα χρηματικό αν θέλετε πρόσωπο, αυτά τα 6 ευρώ οικονομίε. Άρα υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θα μπορούσαν λοιπόν και οι κυβερνήσει ε, να δώσουν το καλό παράδειγμα. Αν συνδέσουν τις δημόσιες προμήθειες με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο αν μπορείτε στα 243 δισεκατομμύρια. Δεν κατάλαβα ακριβώς ε, η κατανομή πώς γίνεται. Κυβερνήσεις, ε, επιχειρήσεις. Και ένα άλλο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχετε ίσως στοιχεία αν κάποιες χώρες τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιες άλλες και γενικώ πώς έχει κατάσταση. Τέλος, είπατε ε, για το 2015 ένα στόχο του 5%, αλλά για το 2020 τι στόχους έχουμε. Ευχαριστώ. Να ξαναδώσουμε λοιπόν το λόγο στους ομιλητές. Ο κύριος Κατινά Το πρώτο ερώτημα είναι και το πιο δύσκολο. Δυστυχώς δεν έχουμε πλήρη και πιστική διάγνωση τέλο τέλος πάντων μια διάγνωση με την οποία να συμφωνούν όλοι για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εάν είχαμε αυτές τις γνώσεις θα ήταν αυτονόητο πως στις διάφορες ανακοινώσεις μας θα είχαμε επιλέξει την οδά αυτή. Η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι η εξής. Έχουμε εντοπίσει κάποια στοιχεία τα οποία παρακολούν την πρόοδο και θέλουμε σιγά σιγά τους φραγμούς αυτούς να τους άρουμε. Τι θα συμβεί αυτό όμως. Όσο υπάρχουν αυτά τα σημεία εμπλοκή, αυτή η φραγμή, υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορεί να αναπτυχθεί απρόσκοπτα το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγηση. Αν λοιπόν είχαμε ένα μηχανισμό, ιδίω μέσω αυτών των φόρουμ, είτε εθνικών είτε ευρωπαϊκών, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε με σταθερό τρόπο να εντοπίζουμε τους παράγοντες αυτούς που δημιουργούν ε, πρόβλημα και σιγά σιγά να τους εξαλείψουμε. Άπαξ και το πετύχουμε αυτό, νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα δούμε έκρηξη, ε, εκτείναξη των ποσοστών ηλεκτρονικών τιμολογίων. Εγώ ε, θα σας πω ότι έχουμε διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα τι θα γίνει στο μέλλον μέχρι το 2018 ε, για παράδειγμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις θέσεις προτεραιότητες, για τα κοινά πρότυπα, common standards, νομίζω για λόγους ε, σαφήνειας θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση τη σημειασιολογία αφενός και τεχνολογία αφετέρου. Στο τέταρτο πυλώνα έχουμε εντοπίσει το μοντέλο UNICEF Act που είναι σημασιολογικό ε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εκεί τυποποιούμε και εξηγούμε τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, σε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Υπάρχει πολύ ξεκάθαρη σειρά και έτσι μπορεί κανείς να ξέρει σαφώς ότι εδώ πρόκειται για το ονοματεπώνυμο, για την τιμή και ούτω καθεξής. Και αυτό δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε το στάδιο αυτό. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί λοιπόν μαζί με το UNCFACT θα πρέπει να ε, συνεργαστούν και έχει υπάρξει και αναδιάρθρωση γιατί υπήρξαν ζητήματα γραφειοκρατικά δυστυχώς όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Πάντως τώρα ε, πλέον η οργάνωση έχει, ε, είναι επιχειρησιακή και μπορεί να ξεκινήσει την εργασία της αυτό το σημασιολογικό αν θέλετε επίπεδο για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτού του ενιαίου μεσολογικού μοντέλου. Για τα τεχνολογικά τώρα, να μην ε, αυταπατώμεθα. Δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ένα ενιαίο σύστημα. Υπάρχουν πολλά συστήματα. Αυτό δεν είναι όμως και δραματικό. Από τη στιγμή που θα ψηφιοποιηθούν τα πάντα θα μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα διεπαφής, interface που σιγά σιγά θα μπορεί να εξασφαλίζει αυτή τη διαλειτουργικότητα που επιθυμούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες προμήθειες, τις συμβάσεις, Νομίζω, προσωπική άποψη, είναι ότι οι δημόσιε προμήθειε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ώστε ο επαγγελματικό κόσμο, ο επιχειρηματικό κόσμο να στραφεί περισσότερο προ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ιδίω στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ στις τέσσερις ομάδες εργασίας, μία από αυτές ε, θέλει ε, να εντοπίσει κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Αυτή είναι η δουλειά της. Ξέρουμε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει αποφάσεις που καθιστούν υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε κάθε συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση, ιδίω για τα procurement, για τις συμβάσεις. Φυσικά, του χρόνου θα εργαστούμε σε συνεργασία με το φόρουμ και τον πρόεδρο που ορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ τον πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ, θα πρέπει λοιπόν να μας διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Και αν πράγματι είμαστε πεπισμένοι ότι οι δημόσιες προμήθειες μπορούν να έχουν θεμελιώδη ρόλο για να τραβήξουν κόσμο προς ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτό. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή σκέφτεται να μην προβεί να δώσει υποχρεωτικό χαρακτήρα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ε, στη δημόσια διοίκηση αλλά το συζητούμε ακόμη και θα εξαρτηθούν πολλά και από τις συστάσεις του φόρουμ. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μελέτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για το ερώτημα, διότι βλέπουμε πολύ καλά που έγκυται το πρόβλημα, η δυσκολία. Αν κάποιος είναι λογικός, ε, νομίζω ότι εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τόσο μεγάλης είναι οι οικονομία που οπωσδήποτε οι πρέπει όλες να στραφούν στην ηλεκτρονική τιμολογία. Γιατί δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν γιατί παραμένουν αβεβαιότητες, άφησε. Υπάρχει και ένα πολιτιστικό ε, πρόβλημα, η αντίσταση στην αλλαγή. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε την απόφαση αντί για τις επιχειρήσεις. Σίγουρα αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, εξαλείφουμε σταδιακά τα εμπόδια, αλλά θα πρέπει οι ίδιες οι επιχειρήσεις ε, να πιστούν και άρα εδώ έχουμε το σκέλος της επίδειξης και τα φόρουμ είναι αυτά που θα έχουν την το ρόλο, να δώσουν απτά στοιχεία για να δείξουν ότι το πέρασμα, η μετάβαση στα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι κάτι που μπορούν να το διαχειριστούν οι επιχειρήσει, δεν είναι ε, καθόλου τοπικό και ανεδαφικό, είναι κάτι πάρα πολύ συμφέρον ε, αντιθέτω. Και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι τα φόρμα μπορούν να κάνουν πολλά. Για το ερώτημα του κυρίου Κέλλη θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Ναι, κύριε Κατινά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να πω ως συμπλήρωμα σε απαντήσει του κύριου Κατινά είναι το εξής. 6 ευρώ ανατιμολόγιο ή 30 ευρώ ανατιμολόγια εξαρτάται από τις μελέτες αλλά και από το εύρος ε, της όλης διαδικασίας. Τέλος πάντων, εξαρτάται από τη σκοπιά το εξτάζει κανείς. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ένα στους 10 προμηθευτές μόνο στέλνει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, δεν μπορεί το όφελος να είναι μεγάλο, αυτό είναι προφανές. Ναι, μεν λοιπόν υπάρχει τεχνολογία και υπάρχει και η σχετική νομοθεσία που το επιτρέπει, υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα ακόμη τα οποία υφίστανται. Και έχουμε και το θέμα του ΦΠΑ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, αν ένα στους δέκα, παραλαμβάνω, μόνο προμηθευτή στέλνει ε, ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, γιατί να μπω στον κόπο να έχω παράλληλα δύο συστήματα, ε, το έντυπο και το ηλεκτρονικό. Άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο όγκο πρώτα απ' όλα και να έχουμε αυτή την ανάγκη το καθολικό τιμολόγιο, το πρότυπο. Οι προμηθευτές, 45 με 65% ανάλογα με το κράτος μέλος, κάνουν τις ε, συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, έχουν μάλλον συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, άρα εδώ έχουμε μεγάλο δυναμικό και αν θέλει οι κυβερνήσει να ζητήσουν από αυτές τις εταιρείε να στέλνουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, θα πρέπει να τους δώσουν και κάποιες προδιαγραφές τυποποιημένες. Ανάλογα με τα διάφορα πρότυπα που έχουμε, το σύφακτι άλλα και... Αν υλοποιήσουν και εφαρμόσουν και κάποιες συγκεκριμένες μεθόδους συμμόρφωσης, μαζί με αυτές τις προδιαγραφές και τις οδηγίες που θα δώσουν, ώστε να μπορούν ε, οι εταιρείε να εφαρμόσουν τα σχετικά, δίνοντας δε δηλαδή το καλό παράδειγμα. Οι διοικήσει, οι κυβερνήσει μπορούν να γίνουν κάποια θετικά πράγματα. Αύξηση όγκου λοιπόν, ε, η ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των προτύπων και η παροχή βέλτιστων πρακτικών για να υπάρχει συμμόρφωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσω το καλό παράδειγμα, αναλαμβάνω, οι κυβερνήσεις, οι διοικήσεις των κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιαζόμαστε και λυπώ γι' αυτό, λυπούμε γι' αυτό, συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν πολύ χρήσιμο όλα όσα μας είπατε. Περνάμε ήδη στον τρίτο γύρο συζητήσεων. fahren fort und begrüßen Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την ε, κυρία Ανδριανή Φέρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαλειτουργικών Συστημάτων και σας δίνω αμέσως λοιπόν το λόγο να ξεκινήσετε εσείς. Thank you very much. I... Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Ανδριανή Φόρτη και είμαι εδώ εκ μέρους του κυρίου Τόμας Βίνια, ο οποίος ζητά συγγνώμη που δεν κατόρθωσε να είναι παρόν. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Τικάου που μας κάλεσε να συμμετάσχουμε σε αυτή την σύντομη ακρόαση που οργανώνει η Επιτροπή σας. Θα ήθελα να πω ότι κατά τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δημόσιες διοικήσεις έχουν καταβάλει προσπάθειες για να διευρύνουν τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μέσα στο ίδιο το κράτος μέλος, αλλά και διασυνοριακά, που είναι το βασικό μας θέμα συζήτησης. Για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να παρέχουν διαμεθοριακές υπηρεσίες, ε, είναι βασικό στοιχείο η διαλειτουργικότητα είναι βασικό για να μπορέσουμε να λύσουμε τα μέγιστα ωφέλη από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με βάση τις προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την τυποποίηση από τον Ιούνιο πέρυσι, το Κοινοβούλιο έχει συνεισφέρει για τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο κανονισμός αυτός θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα για τη δημόσια διοίκηση. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ταχεία έγκριση της πρότασης αναθεώρησης για να επωφεληθούμε από τη διαλειτουργικότητα με βάση τα ανοιχτά πρότυπα. Η δική μου πρόταση θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της δικής μας συζήτησης. Πρώτον, η σημασία της διαλειτουργικότητας και τα διάφορα νομοθετικά κείμενα που την υποστηρίζουν. Δεύτερον, υπάρχει σαφής ανάγκη για ανοιχτά πρότυπα για να διευκολύνουμε την επιλογή των αγοραστών και το κλείδωμα συγκεκριμένων προτύπων και τρίτον το πακέτο μεταρρύθμισης των προτύπων θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα πρότυπα στις δημόσιες προμήθειες σε θέματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Και εδώ έχουμε και το θέμα των τριών βασικών φορέων Υπάρχουν πολλά έγγραφα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα και που προσπαθούν να προωθήσουν σε γενικέ γραμμέ την διαλειτουργικότητα. Ένα παράδειγμα είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής εδώ και ένα χρόνο για τη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη και το αναθεωρημένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας ε, που δημοσιεύθηκε στις 16-12 του 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της διαλειτουργικότητας κατά την παροχή διαμεθοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κατά παρόμοιο τρόπο η διαλειτουργικότητα έχει κεντρικό ρόλο στην στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη που εγκρίθηκε το Μάιο του 2010. Μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στρατηγική του 2020. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ψηφιακό θεματολόγιο μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον έχουμε διαλειτουργικότητα με βάση πρότυπα και ανοιχτέ πλατφόρμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξετάσει και πολιτικέ και νομοθεσία υπέρ τη διαλειτουργικότητα από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90. Η διαλειτουργικότητα βρισκόταν στην καρδιά των συζητήσεων σχετικά ε, με την οδηγία για το ε, copyright. Υπήρχαν πολλές διατάξεις ε, που δείχνουν την νομοθετική πολιτική που θέλει να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα επίσης βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης της Microsoft και η, γενική, απόφαση του δικαστηρίου το 2007 ζητάει από την ε, Microsoft να δώσει πληροφορίες για διαλειτουργικότητα και αυτό υπενθύμησε το σημαντικό ρόλο παίζουν οι αρχές ανταγωνισμού κατά της κατάχρησης μονοπωλιακής θέσης. Τέλος, η διαλειτουργικότητα βρίσκεται πίσω από την πρόταση μεταρρύθμισης ε, της ε, τυποποίησης που κατέθεσε η Επιτροπή τον Ιούνιο σχετικά με την βελτίωση της τυποποίησης και τη μείωση του κόστους για τις αρχές και τις δημόσιες προμήθειες, ενώ παράλληλα προωθείται η διαλειτουργικότητα. Ας συζητήσουμε τώρα το θέμα λίγο περισσότερο για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Η δυνατότητα ελεύθερης διασύνδεσης και επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας πληροφορικής είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τα άτομα, για τις δημόσιες διοικήσεις, για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η δυνατότητα διασύνδεσης βασίζεται στην ομαλή διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων. Διαλειτουργικότητα λοιπόν σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστού μπορεί να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίε με άλλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και θα μπορούν τις ίδιες πληροφορίες να τις χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα. Η ευρεία διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλών συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον βασίζονται ε, σε συστήματα διαπαθής που θεσπίζουν σαφείς κανόνες επικοινωνίας. Ορισμένα πρότυπα επικοινωνία είναι ανοιχτά, άλλα όμω είναι περιοριστικά και κλειστά και δεν επιτρέπουν το βέλτιστο επίπεδο διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα για, τεχνολο... καταναλωτέ και για επιχειρήσει και επομένω έχουμε ε, έλλειψη διαλειτουργικότητα. Θέλουμε κοινά πρότυπα για να ε, μπορούμε να έχουμε ε, επικοινωνία και μεταξύ πολιτών και μεταξύ καταναλωτών, ώστε οι πολιτές να μπορούν να συνδυάζουν τα προϊόντα τους με άλλους πολιτές και οι καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, τα προϊόντα ελεύθερα. Ε, σε ένα κλειστό περιβάλλον υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τα πρότυπα που μπορούν να εφαρμόσουν οι πολιτές και περιορίζεται η επιλογή των καταναλωτών. Αυτό μπορεί να σημαίνει έλλειψη πρόσβασης, επαχθή ευθύς όρους πρόσβασης και τεχνικούς φραγμούς. Από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι ένας ανοιχτός κόσμος είναι ο κόσμος συνεχούς καινοτομία, πολλών ευκαιριών και μεγάλης επιλογής για τους καταναλωτές. Από την εμπειρία μας επίσης βλέπουμε ότι όταν έχουμε ένα κλειστό σύστημα δεν έχουμε το ίδιο, τον ίδιο βαθμό καινοτομία και περιορίζεται η επιλογή των καταναλωτών θέλουμε οι πολίτες να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τις δημόσιες διοικήσεις απρόσκοπτα και να μην κλείνονται, να μην κλειδώνονται οι καταναλωτές σε τεχνολογίες που παρέχονται από ένα και μόνο πάροχο. Αυτοί είναι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν εφόσον πληρούνται ορισμένοι βασικοί στόχοι για, τη δημόσια, για τις δημόσιες προμήθειες προϊόντων, τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Η συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλά για μη διακριτική μεταχείριση και αυτό πρέπει να ισχύει σε κάθε διαδικασία δημόσιων συμβάσεων που επηρεάζει το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στι δημόσιε συμβάσει. Επιπλέον, οι τεχνικέ προδιαγραφέ στις δημόσιε συμβάσει πρέπει να δίνουν ίση πρόσβαση στου διαγωνιζομένους και να μην δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στο άνοιγμα δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Και οι αναθέτουσες αρχέ δεν θα πρέπει να συντάσσουν τι τεχνικέ του προδιαγραφές κατά τρόπον ώστε να αποκλείουν προϊόντα τα οποία δεν πληρούν κάποιε συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Το τωρινό πλαίσιο για τι δημόσίε συμβάσει απαιτεί από τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτω ώστε να χρησιμοποιούν πρότυπα αναγνωρισμένα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την βελτίωση της διαλειτουργικότητα πρέπει να ισχύει η μεταχείριση προς τους πολιτές, να ισχύει η διαφανής μεταχείριση, να μην συντάσσονται τεχνικές προδιαγραφές κατά τρόπον ώστε να αποκλείονται προϊόντα που πληρούν μόνο συγκεκριμένε προδιαγραφές και τέλος δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη μάρκα ή μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις. Και αυτά είναι σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ισχύει η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νομοθετικέ προτάσει για την μεταρρύθμιση τη τυποποίηση που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο και που βρίσκονται τώρα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύουν το ισχύον καθεστώ, τονίζοντα την ανάγκη οι δημόσιε αρχέ να χρησιμοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα σχετικά πρότυπα σχετικά με την προμήθεια λογισμικού και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιλέγονται πρότυπα τα οποία να μπορούν να εφαρμόσουν όλοι οι προμηθευτές για να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός και να μην υπάρχει ο κίνδυνος lock-in εγκλωβισμού. Θέλουμε να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και διαφάνεια και θα πρέπει να ισχύουν οι αρχές της ουδετερότητας και της σταθερότητας και τα πρώτη που, που αναπτύσσονται από φόρουμ και συμπράξεις ε, θα πρέπει επίσης ελεύθερα να συμμετέχουν. Με βάση όλα τα ανωτέρω και για να επιτύχουμε δίκαιο ανταγωνισμό και αξιοκρατία, είναι απαραίτητο οι δημόσιες αρχές να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της του Ιουνίου του 2011 μιλά ιδιαίτερα για την αναγνώριση των προϊόντων φόρουμ και συμπράξεων που πρέπει να βρίσκονται σε ίση βάση με πρότυπα από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και αναγνωρίζονται τα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ξέρετε, οι διερμηνείς έχουν λίγο πρόβλημα με την ταχύτητά σας, λέει ο Πρόεδρος. Αν μπορούσατε να διαβάζετε λίγο πιο αργά θα ήταν καλύτερα. Ιδίω όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, έχει μεγάλη σημασία τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία που θα χρησιμοποιούνται από τι δημόσιε αρχέ να δίδονται με τρόπο δίκαιο που δεν θα ασκεί διακριτική μεταχείριση και θα συμπεριλαμβάνεται και άδεια βασικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ε, χωρίς περιορισμούς. Αυτή η προσέγγιση έχει ε, υιοθετηθεί τηρώντας τις ε, αρχές της δίκαιης μεταχείρισης. Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί αυτή την προσέγγιση και είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να ενστερνιστούν αυτές τις αρχές και να τις υλοποιήσουν ώστε να καταλήξουν στο στόχο μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να τονίσουμε ότι η υλοποίηση των αρχών του ανοιχτού χαρακτήρα από τα κράτη-μέλη και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας θα είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στα προϊόντα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν ανοιχτά πρότυπα και οι κανόνες ε, πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να παρέχονται είτε από ανοιχτά προϊόντα είτε από προϊόντα που διέπονται από κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως στο πλαίσιο της συζήτησης για τα θέματα τυποποίησης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αυτό έχει ε, μεγάλη σημασία για να προωθήσουμε τη διαλειτουργικότητα και να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών και θα πρέπει να γίνει κοινοτικό δίκαιο αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς. Thank you, Ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν, πώς μπορεί να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προσπάθειες για την τυποποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με θετικό τρόπο και δεν εμποδίζουν την καινοτομία στις ε, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και δεύτερον, ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο προτύπων που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή προκειμένου να αναπτύξουμε πανευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες και πώς μπορεί να αποφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υπερβολικά συγκεκριμένη. Ευχαριστώ. Danke sehr, Frau Ferti. Vielleicht können Sie das σας ευχαριστούμε. Κυρία Φέρτη, θέλετε να απαντήσετε. Of course. Um, ευχαριστώ. Καταρχήν, πιστεύω, όπως είπα και στην ομιλία μου, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν περισσότερη διαλειτουργικότητα και η διαλειτουργικότητα είναι πολύ σημαντική για την πρόθεση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους λόγους ε, που βρισκόμαστε εδώ είναι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποφέρει από έλλειψη διαλειτουργικότητας και φυσικά αυτό αποτελεί και σημαντικό εμποδίο στην ε, καινοτομία τι τελευταίε δύο δεκαετίε. Αυτό για την πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, για το ελάχιστο επίπεδο προτύπων και να μην είναι υπερβολικά συγκεκριμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω βάσει των νομικών μου γνώσεων και όχι των τεχνικών γνώσεων μου. Νομίζω ότι οι προτάσεις έτσι όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο παρέχουν αρκετά λεπτομερείς προδιαγραφές αλλά και γενικές προδιαγραφές προκειμένου να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο για το πώς πρέπει να θετούνται τα πρότυπα για την αποφυγή της υπερβολικής εξειδικευσής. Δεν ξέρω αν απαντώ στην ερώτησή σας, αν θέλετε περαιτέρω διευκρινής. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αν συμφωνείτε θα δώσω και πάλι το λόγο στη συνάδελφο Τικάου και από ό,τι μου λένε καθυστερεί ίσω ο επόμενος ομιλητής. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Τικάου για να κάνει την σύνοψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους ε, που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες ε, που μας παρουσίασαν τις δικές τους απόψεις και τις συστάσεις τους. Σχετικά με το τι γίνεται και το τι θα πρέπει να γίνει στα κράτη-μέλη, αλλά και στις διάφορες εταιρείε αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το τελικό πόρισμα είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει όλοι να συνεργαστούμε να εργαστούμε από κοινού. Ναι, χρειαζόμαστε κάποιο είδους τυποποίησης ε, των δεδομένων. Ε, είναι πολύ σημαντικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποτελεί και ένα στοιχείο που πραγματικά θα ήταν χρήσιμο σε όλες τις ε, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και η ηλεκτρονική τιμολόγηση ιδανικά δεν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με τα συστήματα δημοσίων συμβάσεων, δημοσίων προμηθειών, αλλά θα πρέπει να συνδέεται και με τα εμπορικά μητρώα, με όλα τα μητροεπιχειρήσεων ε, που καταβάλουν ΦΠΑ και αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη σε οριζόντιο επίπεδο αν θέλουμε να πετύχουμε την διαλειτουργικότητα των διάφορων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι πρόοδο θα σημειωθεί στην αμοιβή αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα βρισκόμαστε εν μέσω μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ ηλεκτρονική υπογραφή και επαλήθευση τη, ε, authentication. Ένα ε, πολύ σημαντικό αριθμό εμπειρογνωμόνων θεωρούν θεωρεί ότι τα δημόσια συστήματα υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία και η προσέγγιση αυτή είναι παρόμοια με τη σημερινή προσέγγιση για τις υπογραφές. Η, οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές ορίζει την ηλεκτρονική υπογραφή ως μια συλλογή ηλεκτρονικών δεδομένων που επισυνάπτονται ή συνδέονται λογικά με άλλα δεδομένα και που χρησιμεύουν ε, για την ε, επαλήθευση. Έχουμε δηλαδή μια νομική βάση αν θέλουμε να συνδέσουμε την επαλήθευση με την ηλεκτρονική υπογραφή. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των ε, δύο αυτών functionalities, των δύο αυτών λειτουργιών. Πρακτικά, οποιαδήποτε υπογραφή θα αποτελεί και ένα μηχανισμό επαλήθευσης, συνθηκές σε έναν βαθμό, αλλά για τους ε, σκοπούς της ηλεκτρονικής επιγραφής η επαλήθευση αυτή που αναφέρεται στην οδηγία θα μπορούσε να παραβεί στην επαλήθευση των δεδομένων και όχι απαραίτητα στην ε, επαλήθευση, στην ταυτοποίηση της οντότητας που κρύβεται πίσω από αυτή. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι οποιαδήποτε διαδικασία που διασφαλίζει μόνο την ε, επαλήθευση της ταυτότητας της οντότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν μπορεί να έχει αυτό το στάτους και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι πολλές χώρες που έχουν ε, εφαρμόσει διάφορες μεθόδους ε, για αυτή την επαλήθευση των οντοτήτων, θετικές συνοφέτων, βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Και εκεί όπου η μέθοδο αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο φιλικές προς το χρήστη, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο ασφαλής. Το επίπεδο ασφάλεια είναι χαμηλότερο. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή αλλά και η ηλεκτρονική ταυτότητα αντικατοπτρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο στο μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για το ότι ε, η εθνική εναρμόνιση των λειτουργιών ε, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή στο εσωτερικό, στα πλαίσια των ε, διάφορων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικύλουν μεταξύ των διάφορων χωρών. Υπάρχουν μόνο κάποιες χώρες που έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένε διατάξει στην ηλεκτρονική υπογραφή, ενώ πολλέ χώρε επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενό εθνικού πλαισίου για την ηλεκτρονική επιγραφή και λιγότερο επικεντρώνονται στις ε, διασυνοριακές πτυχέ της διαλειτουργικότητας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι για την ανάπτυξη των εφαρμογών που βασίζονται σε ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών, προκειμένου να κυρώνονται οι υπογραφέ αυτές, να επικυρώνονται, θα είναι το πιο σημαντικό να έχουμε μία ομοσπονδία αρχών επαλήθευση αρχών επικύρωσης. Η έννοια βασίζεται στο One Stop Stop, στη μία και μόνη θηρίδα επικύρωσης από τις αρχές αυτέ Και αυτή, η επικύρωση, αυτή την επικύρωση ε, αυτή η επικοινωνία πείτε από τις εθνικέ αρχές στα κράτη-μέλη και έτσι λοιπόν θα διασφαλίσουμε την αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Και θέλω να αναφέρω και το εξή ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να είναι διαλειτουργικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα και την ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά και σε ό,τι αφορά τις δημοσίες υποδομές τους. Σύμφωνα με τις μελέτες της Κομισιόν, πέντε κρατή-μέλη σήμερα διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο γιατί έχουν διασφαλίσει πλήρη διαλειτουργικότητα και έχουν φτάσει στο ψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας, ε, σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών οικονομικής διακυβέρνηση Αυστρία, Μάλτα, ε, Πορτογαλία, Σουηδία και Σλοβενία. Αλλά μιλάμε μόνο για πέντε παραδείγματα του πόσο αποτελεσματικά και διαλειτουργικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα από την Κομισιόν, το ΠΕΠΟΛ, το οποίο είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ένα διασενοριακό σύστημα για τις δημόσιες προμήθειες που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική οδό, το Project Brita. Και Θέλω να πω ότι και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναφέρομαι εδώ στο νομικό πλαίσιο, δηλαδή τα πρότυπα, την υποδομή, τις εφαρμογές και τη διαχείριση αυτού. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλουμε να φτάσουμε στη διαλειτουργικότητα και αν θέλουμε να παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν ε, υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα ούτε καν να ε, δούμε τις ε, δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται δια της ηλεκτρονικής οδού. Δεν μιλώ ε, λοιπόν εδώ για καμία διασυνορική υπηρεσία, αλλά δυστυχώς και στο εσωτερικό ορισμένων κρατών μελών οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι διαλειτουργικές. Σημαντική είναι και η ασφάλεια όταν μιλάμε για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να σας πω ότι η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εναλλακτικών κατά, την, κατά το έτοιμά μου ξεκίνησε μια μελέτη που αφορά την ασφάλεια των ε, συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος ε, και φυσικά Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν τις ε, συνεδριάσεις της ΤΟΑ και αν ε, θέλετε θα σας στηρώ ενήμερους για τις εξελίξεις ε, και μπορείτε να συμμετέχετε και ενεργά στο όλο εγχείρημα αν το επιθυμείτε. Και καθώς μιλούμε για ασφάλεια και για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα ήθελα να σας πω ότι είδα κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν ε, τις επιθέσεις κατά των συστημάτων ε, ηλεκτρονικών ε, δημόσιων προμηθειών. 53,2% Είχαμε λοιπόν 53 μεσές σοβαρές, 40% χαμηλή σοβαρότητας και 2, 5% ήταν πολύ σοβαρές επιθέσεις. Ε, όταν μιλάμε για πολύ σοβαρές επιθέσεις σημαίνει ότι προσπαθούσαν ε, να ε, πάρουν τα δικαιώματα του διαχειριστή, τα δικαιώματα ορισμένων χρηστών. Είχαμε επιθέσεις κατά εφαρμογών στο διαδίκτυο, web applications, επίσης σε επίπεδο πρωτοκόλλων. Είχαμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα είδη των επιθέσεων ε, για το πρωτόκολλο UDP 20%. 34,7% και 45,89%. και αν ε, θέλουμε συστήματα που είναι πραγματικά διαλειτουργικά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση για να πετύχουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά χρησιμοποιούμαστε και σε επίπεδο ασφάλειας ε, και σε επίπεδο υπηρεσιών επικοινωνίας αλλά και σε επίπεδο εφαρμογών που χρειαζόμαστε που χρειάζονται για να πετύχουμε αυτή την διαλειτουργικότητα. Και θα κλείσω λέγοντας όταν μιλάμε για την ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να δούμε και την στάση των χρηστών. Πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι φιλικά προς το χρήστη. Τα πρότυπα είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να εξελίψουμε την πολλαπλή αποθήκευση δύο δεδομένων στο ίδιο σύστημα επίσης και το φορμάτι των δεδομένων είναι πολύ σημαντικό και σχετικά πρόσφατα είδαμε την υιοθέτηση μιας δεσμής μέτρων που αφορούν τα ανοιχτά δεδομένα. Πρακτικά αυτή η δεσμή μέτρων ε, θα αλλάξει την οδηγία που αφορά τη χρήση των αποθηκευμένων ε, δεδομένων από τους δημόσιους φορείς, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει προσβασιμότητα στα δεδομένα αυτά και ότι είναι συμβατικά αυτά τα δεδομένα, συμβατά αυτά τα δεδομένα, με συγχωρείτε. όλα αυτά τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφοριών των διάφορων δημόσιων φορέων θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα, θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα και θα πρέπει να είναι σε ένα μορφότυπο που να είναι συμβατό με τις μελλοντικέ τεχνολογικές εξελίξεις. Και Συμπερασματικά υπογραμμίζω το πόσο σημαντική είναι η μηδένα αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Πόσο σημαντικό είναι το νομοθετικό πακέτο που θα έχουμε του χρόνου σε ό,τι αφορά τις αλλαγές ε, στην οδηγία που ρυθμίζει τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Και επίσης και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, ως προς την ηλεκτρονική ταυτότητα. Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική υπογραφή πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρχών Επικύρωσης. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε την αμοιβή αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Πιστεύω ότι έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι. Είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους πόρους για τα πιλωτικά προγράμματα και για τα προγράμματα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα των διάφορων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν και αυτά αρκετά κονδύλια για την εφαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο. Και τα πρότυπα είναι ουσιαστικά αλλά και ασφάλεια. Ορισμένες πρωτοβουλίες μπορούν να μας βοηθήσουν ε, να πείσουμε τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις ε, για να υιοθετήσουν αποτελεσματικές λύσεις όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση ή η πρόσβαση και χρήση διάφορων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ελπίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Ευχαριστώ όλους τους ε, προσκεκλημένους και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που περιβρέθησαν εδώ σήμερα Φυσικά να σας πω ότι είναι να λάβω τις τροπολογίες των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και κλείνουμε τη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών σε πέντε λεπτά.